Να περάσουμε τώρα απευθείας ε, στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Δήλωση και πάλι της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Πυρηνική Απειλή και Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα. Κύριε Αστόν, έχετε το λόγο. Η Βόρεια Κορέα είναι η πιο απομονωμένη χώρα στον κόσμο και η πιο εχθρική στους γείτονές της. Ο λαός της, πέραν μιας μικρής ελίτ, ε, ε, ζουν καθημερινές στερήσεις. Ε, δεν υπάρχουν επαρκή τρόφιμα και αυτό σημαίνει ότι εξαρτώνται συνεχώς από διεθνείς χορηγούς. Παρά το γεγονός ότι έχουμε μια τρίτη γενεά ηγετών, υπάρχουν κάποιες αποτυχημένε απόπειρε οικονομική μεταρρύθμισης, δεν διαπιστώνεται ότι υπάρχουν κάποιες βελτιώσει ενώ ταυτόχρονα ο, ο λαός πάσχει, το καθεστώς ε, καταξοδεύει πόρους για ε, μεγάλους ε, αμυντικούς ε, εξοπλισμούς ε, και πολύ τεχνολογικά εξελιγμένα επιθετικά όπλα. Οι συνομιλίες ε, των έξι ε, πλευρών δεν έχουν αποτελέσματα και φαίνεται ότι υπάρχει ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. είδαμε μία εκτόξευση πυράβλου το Δεκέμβριο και μία πυρονική δικημή το Φεβρουάριο και αυτό φυσικά οδήγησε σε μία σειρά από απειλές όταν η διεθνής κοινότητα διαμαρτυρήθηκε. Αυτό αποτελούν ε, κατάφορη πρόκληση στο καθεστώς μη διάδοσης όπλων και μια σοβαρή απειλή στην ειρήνη. Εμείς ταυτόχρονα και οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, συνεχώς ε, διευκρινίζουμε ότι αν η Βόρεια Κορέα ξεκινήσει να, με τις προσπάθειες να κάνει μια ουσιαστική αλλαγή θα τη βοηθήσουμε. Εγώ αναφέρθηκα στα σημεία τα οποία μας ανησυχούν για την Βόρεια Κορέα με τους ομολόγους μου από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών. Κυρίως ε, ζητήσαμε από την Κίνα να ασκήσει πιέσεις στο καθεστώς της Πιονγιάνγκ και αυτό φυσικά θα βρίσκεται στις προτεραιότητές μου όταν θα επισκεφθώ την Κίνα τον επόμενο μήνα για την ανάπτυξη των σχέσεων με τη νέα ηγεσία. Ε, είδαμε σε επαφέ και με την Νότια Κορέα και η κυβέρνηση της Νότια Κορέα ε, δήλωσε ότι είναι διατεθειμένη να ξεκινήσει ε, συζητήσεις και αυτό φυσικά ε, έρχεται να προσθεθεί στα όσα λέει η Κίνα προσφάτως ε, για το διάλογο. Θέλουμε να αποστείλουμε σαφή μηνύματα προς την Βόρεια Κορέα και να του τονίσουμε ότι δεν θα δεχτούμε συνεχείς παραβιάσεις στο καθεστώ μη διάδοσης όπλων. Το ψήφισμα 2094 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συμφώνησε στις 7 Ματρίου ε, να επιβάλλει μια σειρά από νέα περιοριστικά μέτρα, κυρίως στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Ε, διευκρινίζει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα αναλάβει περαιτέρω δράση αν συνεχίσει να καταπατά του διεθνού κανόνε η Βόρεια Κορέα. Ε, χαιρετίζω τι ε, διπλωματικέ προσπάθειε των Ηνωμένων Πολιτειών και τη Κίνα και τη Ρωσία, ε, που οδήγησαν στην ενότητα στο Συμβούλιο Ασφαλείας και ενδιαφέρονται και για το τι θα συμβεί με τους γείτονες. Ε, υποστηρίζουμε τις συνομιλίες ε, των έξι πλευρών ε, τα τελευταία χρόνια και μας ενδιαφέρει να υπάρχει ειρήνη διότι υπάρχουν και οικονομικά συμφέροντα και θέματα ασφυλίας στην περιοχή. Υποστηρίξαμε και το καθεστώς των Ηνωμένων Εθνών και τη διάφορα ψηφίσματα μετά από τις διάφορες πυρηνικές δοκιμές που είχαμε και το 2006 και το 2009 και πιο πρόσφατα το Δεκέμβριο του 2012 και το Φεβρουάριο του 2013. Θα πρέπει να έχουμε ε, βασικές πτυχές για τον τομέα των βαλιστικών πυράβλων, κάποιες ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές από την ε, Κεντρική Τράπεζα της Βόρειας Κορέας και από διαφόρους ε, Κυβερνητικού φορεί. Είμαστε αποφασισμένοι να αναλάβουμε δράση σε απάντηση στι προκλήσεις. Η πιο πρόσφατη ήταν μια μονομερής δήλωση ότι η ε, εκεχηρία του 1953 είναι άκυρη και ε, την απειλή του Κιμ Γιονκού να εξαφανίσει ένα μικρό νησί της Νότιας Κορέας. Όλες αυτές οι προκλήσεις είναι απαράδεκτες και γι' αυτό ακριβώ στι 18 Φεβρουαρίου το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ανέκρινε ένα ε, ε, νέο, μια νέα δέσμη μέτρων, τα οποία ενισχύουν περαιτέρω τα μέτρα τα οποία εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 22 Ιανουαρίου. Μα ανησυχούν ιδιαίτερα και τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα βοηθήσουμε, θα συμμετέχουμε σε ένα ψήφισμα με την Ιαπωνία στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενέβη για τη δημιουργία μια ανακριτική επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι παραβιάσει του στην Βόρεια Κορία. Το 2011 δώσαμε 10 εκατομμύρια ευρώ για να ανταποκριθούμε σε κατεπίγουσες ε, ανάγκες επισητιστικές ε, μέσω του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων. Ε, η βοήθεια αυτή δόθηκε στις πιο ευάλωτες ομάδες για να βελτιωθεί η διατροφή των παιδιών κάτω των 5 ετών στα ορφανοτροφία, οι έγκες γυναίκες και οι ηλικιωμένοι και οι ανάπηροι. Θα συνεχίσουμε να βοηθούμε τα Ηνωμένα Έθνη στις προσπάθειές τους για να διατηρήσει ενωμένη τη διεθνή κοινότητα και μόνο αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε το καθεστώς μη διάδοση όπλων και να υποστηρίξουμε το λαό της Βόρειας Κορέας. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων τώρα, ο κύριος Έλμαρ Μπρόκ για δύο λεπτά, εξ ονόματος του ΕΛΚ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπατή, εκπρόσωπη και αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σα ευχαριστώ κυρία Άστον για τα όσα μα είπατε εδώ και για τα όσα έχετε επιτύχει τις τελευταίες εβδομάδες η Βόρεια Κορέα. Είναι ένα κράτος το οποίο καταπιέζει τους πολίτες του, επιβάλλει πολλά δεινά σε αυτούς και είναι και επιθετικό κράτος. Είναι ένα κράτος το οποίο φαίνεται να κατασκευάζει πυρηνικά όπλα, να τα δοκιμάζει, να τα συνδυάζει με πρόγραμμα πυραυλικό και ταυτόχρονα καταγγέλει την συμφωνία για τους, ε, εξοπλισμού, για τους του 53, όπως είπατε. Μια συμφωνία η οποία θα μπορούσε να κατασυγάσει τα πνεύματα, ενώ βλέπουμε λοιπόν να συγκεντρώνει στρατεύματα και να οξύνει το κλίμα βρισκό, σημαίνει ότι βρισκόμαστε ενώπιον ενός άμεσου κινδύνου πολέμου και άρα συνθήκων που θα μπορούσαν και μακροπρόθεσμα να ανατρέψουν την εικόνα της περιοχής. Η επιθετικότητα του κράτους αυτού, συνδυασμένη με την πυρηνική του δύναμη, είναι πολύ επικίνδυνη για την περιοχή αυτή. Φυσικά θα μπορούσε κάποιο να προτείνει την ιδέα να εξοπλιστούν με πυρηνικά και άλλα κράτη για να μπορούν να απαντήσουν σε αυτήν την απειλή, αλλά αυτό θα σημαίνει το τέλο του Συμφώνου περί μη διάδοση των πυρηνικών. Και εδώ πρέπει να βάλουμε στην εικόνα και το Ιράν και τη στάση του. Έχουμε λοιπόν μεγάλο κίνδυνο πυρηνικού πολέμου, κίνδυνο που δεν είχαμε μέχρι τώρα ποτέ. Εδώ η Κίνα έχει να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι καλό το ότι μπορέσετε να εξασφαλίσετε τη συνδρομή της Κίνας στις προσπάθειές σας. Μόνο όμως ε, η Κίνα, από την οποία εξαρτάται τόσο ουσιαστικά η Βόρεια Κορέα για πάρα πολλά πράγματα, είναι ε, σε θέση να επηρεάσει την κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να συνομιλήσετε με την Κίνα, να την πείσετε να αλλάξει στάση απέναντι στη Βόρεια Κορέα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκόμες έχει το λόγο. οι απειλές του καθεστώτος Βόρειας Κορέας ε, είναι απαράδεκτες ε, και δεν απευθύνονται μόνο στην Ιαπωνία, την Νότια Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, απειλείται και η συνολική ασφάλεια. γίνεται παραβίαση του συνθήκης μη διάδοση πυρηνικών όπλων, η ανακοχή ε, μεταξύ Βόρειας και Νοτιάς ε, Κορέας και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ε, όλα αυτά θέτουν σε κίνδυνο και την ίδια ασφάλεια της Βόρειας Κορέας. Η οικονομία της Βόρειας Κορέας έχει επικεντρωθεί στα οπλικά συστήματα και οδηγεί σε ακραία φτώχεια το λαό, ο οποίος επίσης πλήττεται από παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προ ψευδή προπαγάνδα, καταπίεση κλπ. Γνωστού του Ε, μπορεί να είναι φεοδαρχική, τρελή ή ε, καταπιεστική η κυβέρνηση, αλλά ε, αυτή τη ε, στιγμή ε, υποστηρίζεται οικονομικά και πολιτικά από την Κίνα και μόνο έτσι στέκεται στα πόδια της. Ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ η Κίνα έχει ευθύνες. Πρέπει να ξεκινήσει ε, από τη γειτονιά της. Δεν είναι δυνατόν. Δεν, δεν είναι δυνατόν να δέχεται ε, τις ε, κυρώσεις του ΟΗΕ, να επιτρέπει να ψηφιστούν και μετά να βοηθάει ε, το καθεστώς του, της Βόρειας Κορέας. Θα πρέπει να βοηθήσει να πιεστεί το καθεστώς της Πιον θα θέλουμε μια ε, ε Κορέα ε, ελεύθερη από πυρηνικά όπλα και με τους λαούς της Βόρειας της Κορέας να ζουν σε ειρήνη. Θα πρέπει να προωθήσουμε τις κυρώσεις εναντίον της Πιον Γιάνγκ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διατηρήσει και να ενισχύσει το διάλογο με το καθεστώς της Βόρειας Κορέας και ενδεχομένως, αν είναι δυνατόν, και με την κοινωνία των πολιτών. Όμως οι πιέσεις θα πρέπει να εστιαστούν κυρίως στην Κίνα. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων για δύο λεπτά ο κύριος Κάτσιν. Κύριε Άστον, αγαπητοί συνάδελφοι, η κρίση ε, στη Χερσόνησο είναι εικονική, αλλά η δικτατορία είναι πραγματική. Τα πρόσφατα γεγονότα στην ε, ε, κορατική Χερσόνησο ε, πηγαίνουν πέραν των προβλέψεών μας και δείχνουν ότι η συμπεριφορά των πολιτικών ε, ηγετών ε, είναι η ίδια είτε στο διεθνές προσκήνιο είτε στο εσωτερικό. Θα πρέπει να υπάρξει δράση, διότι είναι απαράδεκτο και ανεύθυνο να θεωρούμε ότι πρέπει να ε, επανεκπαιδεύσουμε ε, τους πολιτικούς ηθήνοντες. Υπάρχει καταπίεση και βασανισμοί, ε, ακόμα και για τους ίδιους τους πολίτες, με το πρόσχημα της εξωτερικής απειλής της χώρας. Κανείς ε, δεν ε, αποτελεί απειλή, ούτε στρατιωτική, ούτε πολιτική απειλή για τη Βόρεια Κορέα. Η, το κράτος, ε, την οικονομία και τους πολίτες μόνοι τους δημιουργούν τα προβλήματα. Ο νέος ηγέτης της δυναστείας δημιουργεί προβλήματα ακόμα και στον σημαντικότερο εμπορικό της εταίρου και σύμμαχο την Κίνα. είναι ομόφωνη λοιπόν η κατακραυγή. Ο ο Κιμ Τζακούν λέει ότι θέλει πολιτικές μεταρρυθμίσεις, καλύτερο επίπεδο διαβίωσης για τους πολίτες του, αλλά αυτή η επίδειξη ε, στρατιωτικής ισχύως ε, και οι απειλές είναι ένα παιχνίδι πόκερ το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ε, πέσουμε στην παγίδα. Ε, τα θύματα, οι ναύτες οι οποίοι ε, ε, θα πέθαναν στην επίθεση του πυράβλου ε, στην θάλασσα πριν από δύο χρόνια ε, αρκούν και μόνο για το γεγονό ότι πρέπει να λάβουμε μέτρα και θα πρέπει να απαντήσουμε. Θα πρέπει το καθεστώ να αλλάξει στάση και ενώπιον των ίδιων του των πολιτών και να ξεκινήσει η διαδικασία του εκδημοκρατισμού μέσω του σεβασμού των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό ακριβώ είναι πολύ σημαντικό για μα, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και δεν θα πρέπει να υπάρχουν απειλέ ε, και να υπάρχει ε, μια διαφορετική κατάσταση. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Κρόμπερ, για δύο λεπτά. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πράσινοι ενώνουν τη φωνή τους στην καταδίκη των ε, παραβιάσεων ανθρωπινών δικαιωμάτων ε, και των ε, πυρηνικών δοκιμών στην Βόρεια Κορέα και την καλούν να μην συνεχίσει αυτές τις πυρηνικές δοκιμές. Καλούμε την ε, ηγεσία της Βόρειας Κορέας να τηρήσει τις αρχές του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, να επανέλθει στην Συμφωνία περιμιδιάδοση των Πυρηνικών και να υπογράψει το συμπληρωματικό πρωτόκολλο. Πρέπει να εφαρμόσει μορατόριο στις δοκιμές των πυράβλων, να υπογράψει και να κυρώσει την ε, συνθήκη περί πυρηνικών δοκιμών. Λυπούμαστε ωστόσο που το ψήφισμα δεν τοποθετείται περισσότερο όσο πόσο θα, έχουν, πρέπει να κάνουν και τα υπόλοιπα κράτη που διαθέτουν πυρηνικά για να αποτρέψουν πυρηνικά χτυπήματα ή ακόμα χειρότερα πυρηνικό πόλεμο. Τα κράτη που διαθέτουν πυρηνικά, συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να διαρρήξουν το δεσμό μεταξύ του καθεστώτος και του κύρους τους και τη κατοχή των πυρηνικών. Και έτσι λιγότερο ε, λιγότερα κράτη θα επιδιώκουν για να ενισχύσουν τη θέση τους στο παγκόσμιο σκηνικό να αποκτήσουν πυρηνικά όπως η Βορεια Κορέα. Πρέπει τώρα λοιπόν όλες οι χώρες που έχουν προσπογράψει τη συνθήκη περί διάδοση των πυρηνικών να συνεχίσουν την πορεία για τον μη για τον αφοπλισμό, για τη συνέχιση του αφοπλισμού και χαίρομαι ιδιαίτερος που τώρα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει οθετήσει την πολιτική για τους αφοπλισμούς. Πρέπει να αγωνιστούμε λοιπόν για τον πυρηνικό αφοπλισμό και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μιγκάλσκι, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, συζητούμε ένα πολύ σημαντικό θέμα εδώ. Την απουσία δημοκρατικών αρχών, δημοκρατικού καθεστώτος στη Βόρεια Κορέα. Λόγω της οποίας το καθεστώς στη χώρα μπορεί να αποτελέσει σημαντική πρόκληση για την παγκοσμία ειρήνη. Ας μιλισμονούμε τους ίδιους Βορειοκορεάτες που υποφέρουν τα πάνδυνα. Νομίζω πρέπει να τους ονομάσουμε κατοίκους του πιο καταπιεστικού, του πιο κατασταλτικού καθεστώτος στον κόσμο σήμερα. Και σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας πιστεύω ότι πρέπει να μεριμνήσουμε για την διαφύλαξη της ασφάλειας, να αντιμετωπίσουμε τις πυρηνικές δοκιμές και να προστατεύσουμε αυτούς τους πτωχούς Νότιο-Κορεάτες οι οποίοι υποφέρουν λόγω της ε, κυβέρνησής τους και του καθεστώτος στη Βόρεια Κορέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπάφτον δεν είναι εδώ, θα λάβει το λόγο ο κύριος Σόλτς. Ο κύριος Σόλτς από την ΚΟΕ. Κύριε Πρόεδρε, Ε, πριν από δύο χρόνια ένας μεγάλος σεισμός και το τσουνάμι οδήγησε σε πολλά προβλήματα την Ιαπωνία. Ε, η Κορέα συνεχίζει όμως να επιδιώκει το, την πυρηνική την, ε, πυρηνική, τον πυρηνικό εξοπλισμό. Χειροσήμα το Ναγκασάκι, το Τσέρνομπιλ, το Χάρισμπουκ και η Φουκοσίμα πρέπει να είναι πάντα στο μυαλό μας να συζητούμε την ε, Βόρεια Κορέα και την, ε, τους πυρηνικούς εξοπλισμούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να καταστήσει απόλυτα σαφές ότι δεν υπάρχει δικαίωμα για προληπτικά χτυπήματα μέσω πυρηνικών. Κανείς δεν έχει τέτοιο δικαίωμα ούτε λόγω εθνικών συμφερόντων ούτε, στο όνομα του δημοσίου δικαίου, του διεθνούς δικαίου. Και αυτό ισχύει για όλα τα κράτη του κόσμου. Ωστόσο δεν πρέπει να λησμονήσουμε και ότι οι εξελίξεις στη Βόρεια Κορέα έχουν λόγους ιστορικούς, έχουν αίτια πολύ βαθιά ριζωμένα, ρίζες που ξεπερνούν την πεντηκονταετία και δεν μπορούμε να δούμε τις εξελίξεις αυτές αποκομμένες ούτε αποκομμένες βέβαια από την πολιτική κατάσταση και τον χωρισμό της ε, κορεατικής χερσονήσου. Η επίλυση λοιπόν αυτής της ε, ε, σύγκρουσης, αυτής της διαφοράς μπορεί να βρεθεί μέσα σε, περίπλοκες ε, πολιτικές με τη συνδρομή των ΗΠΑ και της Κίνας που θα πρέπει να βοηθήσουν στην αποκλιμάκωση της κατάστασης. Πρέπει να εξασφαλιστούν οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέλιξη προς την ειρήνη και την ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Διακόπτε Πρόεδρος. Δότς, παρακαλώ. Η κυρία Δότς. Οι παράνομε πυρηνικέ δοκιμέ τη Βόρεια Κορέα ε, τον προηγούμενο μήνα αποτελούν σαφή απειλή προ την διεθνή κοινότητα και ε, ασφάλεια και ειρήνη. Και βεβαίω είμαι υπέρ των σκληρών ε, κυρώσεων εισβάλλων τη χώρα, αλλά οι εξελίξει οι λιγότερο ορατέ είναι ακόμη πιο σοβαρέ, γιατί πίσω από αυτή το, το πυρηνικό εξοπλισμό της Κορέας κρύβεται ο υποσυτισμό και ακόμη και η αναγκαστική εργασία των Κορεατών, της, των κατοίκων της Βόρεια Κορέας η οποία καταγράφεται ως ο πιο δύσκολος ε, τόπος στον κόσμο για να ζήσει χριστιανός. Οι χριστιανοί διώκονται εκεί κατά τρόπο απολύτως απαράδεκτο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αξιοποιήσει τη σημερινή συζήτηση για να, προαγάγει την, ε, για να ζητήσει την προαγωγή της ε, ειρήνης, της ασφάλειας, των δικαιωμάτων, ε, της ελευθερίας της θρησκευτική συνείδησης με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουν οι χριστιανοί να έχουν την ελευθερία της συνείδησής τους και στην Κορέα. Ο πρόεδρος κλείνει το μικρόφωνο της ομιλήτριας. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Κέλλα με 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ο Διευθυντής της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών εχθές ενημερώνει ενημέρωσε για δοκιμές διπυρωτικών πυράβλων με πυρηνικές κεφαλές και να ταυτόχρονα το Ιράν φαίνεται να κάνει παιχνίδια για να κερδίσει χρόνο. Η Βόρεια Κορέα αρχίζει να επιδεικνύει πλήρη παραγνώριση των διεθνών της δεσμεύσεων. Αλλά η Βόρεια Κορέα δεν μπορεί να δραμώνει της. Η Κίνα πιστεύω έχει να δραματίσει κρίσιμο ρόλο εδώ. Και ενώ η Κίνα φαίνεται να βρίσκεται σε αμηχανία από τη συμπεριφορά της Βόρειας Κορέας είναι ακόμα ιδεολογικά συνδεδεμένη με το κράτος αυτό ε, λόγω του κομμουνιστικού της κομμουνιστικής τους ιδεολογίας. Και η Κίνα δεν, είναι, δεν ενδιαφέρεται από ό,τι φαίνεται για την κατάρρευση του κορεατικού καθεστώτος, καθεστώτος στη Βόρεια Κορέα. Ένα άλλο ζήτημα βέβαια είναι η συνεργασία μεταξύ Βορειάς Κορέας και Ιράν. Συνεργασία που, είναι προφανώς, αφορά προφανώς την ε, ανάπτυξη, εμφανώς την ανάπτυξη πυράβλων, αλλά κατά πάσα πιθανότητα και πυρηνικών όπλων. Πρέπει λοιπόν να καταδικάσουμε αυτή την ε, αλληλεγγύη μεταξύ αυτών των κρατών και να ζητήσουμε. Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή. Με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να είμαι σκληρός και αυστηρός. Η κυρία Κοπά, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η καταδίκη μα για τις νέες προκλητικές ενέργειες της Pyongyang είναι απερίφραστη. Είναι ωστόσο σημαντικό να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση και να επικρατήσει η λογική τη ειρήνης στην περιοχή. Το καθεστώ της βόρεια Κορέα πρέπει να φροντίσει τι πραγματικέ ανάγκε του λαού που ζει ήδη σε συνθήκες ανθρωπιστική κρίσης, να βελτιώσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να πάψει να επενδύει σε ανώφελα εξοπλιστικά προγράμματα αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα που στέλνει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο με το αυριανό ψήφισμά του. είναι ιδιαίτερα σημαντικό που το κείμενο δεν περιορίζεται μόνο στις ε, πυρηνικές φιλοδοξίες της πιονγκιάνγκ. οι νέες πυρηνικές δοκιμές της βόρειας κορέας και η κατάσταση σε σχέση με το ιράν πρέπει ωστόσο να αποτελέσουν μια αφορμή για να ξανασκεφτούμε τι έχουμε κάνει λάθος σχετικά με τη μη διάδοση των πυρηνικών φοβάμαι ότι όσο επιτρέπεται σε κάποια κράτη να έχουν πυρηνικό οπλοστάσιο είναι δύσκολο να υπάρξει πιστικό επιχείρημα για την απαγόρευση σε άλλα να τα αποκτήσουν. επίσης η τακτική της απομόνωσης και των κυρώσεων δεν έχει δώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. η λέξη κλειδί πρέπει να είναι engagement και όχι απλώς diplomatic isolation. πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να εμπλέξουμε όλες τις πλευρές σε μια προσπάθεια για γενικότερο πυρηνικό αφοπλισμό οφείλουμε να οικοδομήσουμε στι αρχέ του ανθρωπιστικού δικαίου να κάνουμε σαφέ ότι οι απειλέ για πρώτο χτύπημα δεν έχουν κανένα νόημα. μια τέτοια κίνηση είναι αυτοκαταστροφική για την ανθρωπότητα και αυτή η απλή λογική καθιστά παρανοϊκή την ίδια την ύπαρξη πυρηνικών όπλων στον κόσμο. ευχαριστώ. Καλησπέρα σας Κάθη. Ο κύριος Χέφνερ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, την συνάδελφοι. Είναι πολύ επικίνδυνος ο πυρηνικός ο αγώνα για του πυρηνικού εξοπλισμού. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή στην ε, Κορεατική Χερσόνησο. Μην ξεχνάμε ότι η Βόρεια Κορέα είναι μια δικτατορία που επιβάλλει τρόμο, εξάρτηση, ε, απουσία ανεξάρτητης ζωής στους πολίτες της. Δεν πρέπει να λησμονήσουμε ότι υπάρχει επικρατεί ένα κομμουνιστικό καθεστώς χωρίς ελευθερία του λόγου, ελευθεροτυπία, δημοκρατία, τίποτε από όλα αυτά που θα μπορούσαν να αποτελέσουν έκφραση των ανθρώπινων ελευθεριών. Σε νέα διαφορετικές περιοχές ε, καταγράφονται πολυάριθμες ε, ε, επιβουλές προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα, ιδιαίτερα ε, με φόνους, με βασανισμούς εις βάρος πολιτών και υποχρεώνονται και οι γυναίκες ή τα παιδιά τους να παρακολουθούν την ώρα που βασανίζονται. Όλα αυτά καταγράφονται σε μια ανεξάρτητη έκθεση. Αλλά πιστεύω ότι ακόμη μέσα στο Μάρτιο πρέπει η κατάσταση στη Βόρεια Κορέα να διερευνηθεί διεξοδικά και μετά να αναβλάβουμε κάθε δυνατό μέτρο, οτιδήποτε μας επιτρέπει το Δημόσιο Εθνές Δίκαιο. Ευχαριστώ πολύ. Για μισή λεπτό. Ο Αντιπρόεδρος κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν λειτουργούσε πριν το μικρόφωνο μου, τώρα λειτουργεί. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. κύριε Υπατή εκπρόσωπε, πριν από δύο εβδομάδες ήμουνα με την αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 22η ε, διάσκεψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Γενέβη. Και εκεί στη Γενέβη ε, μπορέσαμε να μιλήσουμε με την αρμόδια από την Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και που ήταν και πρόεδρος στο παρελθόν του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Και μας είπε κάποια πράγματα για την τραγική, πραγματικά τραγική κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα. Τη Δευτέρα ε, ένας από τους εισηγητές ε, των Ηνωμένων Εθνών μίλησε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ερευνητική επιτροπή για να δει πώς ακριβώς έχει κατάσταση στα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα και ε, θα εκριθεί κατά πάσα πιθανότητα αυτή η Επιτροπή. Θα πρέπει να λυθεί το ζήτημα, διότι θα μπορέσει να είναι μια σημαντική φωνή αυτή η Επιτροπή, ελπίζω όχι μόνο για τη διεθνή κοινότητα, αλλά και για το καθεστώς της Βόρειας Κορέα. Ε, αυτά τα οποία γίνονται, οι συνεχείς εκτελέσεις, ο φόβος που επικρατεί, το γεγονός ότι στέλνονται άνθρωποι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης απλώς και μόνο διότι διαφαινούν με το καθεστώς ε, της Βόρειας Κορέας. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφο για ένα λεπτό ο κύριος Κουτάς. Ευχαριστώ πρόεδρε επιθετικές δηλώσεις της Βόρειας Κορέας, Κορέας ε, τελευταία κατέληξαν στην καταγγελία της ε, ανακοχής με την Νότιο Κορέα και σε απειλές πυρηνικής επίθεσης. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ανησυχητικά. Η Βόρειος ε, Κορέα θα πρέπει να ηρεμήσει λίγο σε σχέση με τις επιθετικές κουβέντες που εξαπολύει και να ασχοληθεί περισσότερο με το μέλλον και τη μοίρα των πολιτών της που εξαρτώνται άμεσα από την εξωτερική βοήθεια. Η έξοδος από το αδι... σημερινό αδιέξοδο είναι ο διάλογος και η, ειρηνική συμπεριφορά. Θα πρέπει να σταματήσουν και πάλι τους, τις πυρηνικές δοκιμές ε, και ε, να πάψουν να ε, παραβιάζουν τη συνθήκη μη διάδοση πυρηνικών όπλων είναι και συμφέρον τη Κίνα, ω μονίμου μέλου του Συμβουλίου ασφαλεία του ΟΗΕ να πιστεί η Βόρειο Κορέα να βοηθήσει στην σταθεροποίηση περιοχή περιοχής. Η Κίνα θα πρέπει να πείσει την Πιονγκιανγκ να ξαναεπανέλθει ε, στις ε, συνομιλίες, στι εξαμερεί συνομιλίες. Ε, πιστεύω επίση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διατηρήσει κάποια κανάλια επικοινωνία με τη Βόρεια Κορέα. Για ένα λεπτό ο λόγος στην κυρία Σενίτσιν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Βόρειο Κορέα είναι μία από τις χειρότερες σε όλη τον πλανήτη. Συνεχείς εκτελέσεις ακόμα και ανηλίκων, ε, υποχρεωτική εργασία, καταναγκαστικά έργα ε, καταδίωξη θρησκειών, δολοφονίες, ανθρωποκτονίες, ε, απαγωγές κλπ. Οι διεθνείς ε, οργανώσεις που παρακολουθούν την κατάσταση τα καταγγέλνουν όλα αυτά. Και οι κυρώσεις του ΟΗΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν αλλάξει την κατάσταση και πολύ. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε το διάλογο και πρέπει εμείς θα πρέπει επίσης να κρατήσουμε ενιαία στάση εναντί του καθεστώτος της Βόρειας Κορέας. Διότι η κατάσταση ασφαλείας στη Βόρεια Κορέα επηρεάζει την ασφάλεια σε όλο τον πλανήτη. Το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας, για παράδειγμα, ε, είναι πολύ σημαντικό, όπω επίση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι παραβιάσει των ανθρώπινων δικαιωμάτων πρέπει να σταματήσουν. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό ο συνάδελφος Αρλάκη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Άστον. Ε, συμμερίζομαι την ισχυρή καταδίκη των πρόσφατων πυρηνικών απειλών της Βόρειας Κορέας. Είναι πρόκληση σε ό,τι αφορά το καθεστώς ε, της μηδιάς των πυρηνικών όπλων και σημαντική απειλή στην σταθερή ειρήνη της ε, ε, ε, Χερσονήσου της Κορέας. Είναι η κατάλληλη στιγμή να θυμηθούμε ότι Κανένα κράτο δεν θα πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα, ούτε το Ιράν, ούτε η Βόρεια Κορέα. Ε, αλλά ούτε και οι επικριτές τους. Η, η παγκόσμια ασφάλεια δεν μπορεί να διασφαλιστεί από ένα κλαμπ, μια λέσχη πυρηνικών δυνάμεων. Ε, μέχρι να ξεφύγουμε από αυτά τα δύο μετρακίδια σταθμά ε, και να καταστεί παράνομη η κατοχή των πυρικών όπλων, δεν πιστεύω ότι θα κάνουμε σημαντική πρόοδο σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής για αυτό το θέμα για ένα λεπτό, ο κύριος Ζάλα. Συνάδελφοι, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εμπλακεί πιο άμεσα ε, σε αυτό το αδιέξοδο, θα πρέπει να ενισχύσει την πολιτική της ε, παρουσίας στην Νοτιοανατολική Ασία, καταρχήν. Η, ε, η δραστηριότητα μας στη Μιαμάρα το δείχνει ότι αυτό είναι δυνατό. Σε ό,τι αφορά την πυρηνική κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεισφέρει, για παράδειγμα, μέσω της χρήσης της ε, στρατηγικής συμμαχίας με τη Ρωσία και την Κίνα. Η θέση της ε, Κίνας ό,τι αφορά τη Βόρεια Κορέα θα είναι αποφασιστική σημασία. Αλλά και η θέση της Ρωσίας θα είναι εξίσου σημαντική. Θα πρέπει να εμπλακούν και οι δύο αυτές μεγάλες δυνάμεις. Ε, και είναι δύσκολο. Εκεί η ευρωπαϊκή διπλωματική δράση έχει μεγάλο πεδίο δράση. Περνάμε στην διαδικασία του Catch the Eye. όσο μας επιτρέπει ο χρόνος. Ε, στο ένα λεπτό θα σας σταματάω. Ο λόγος στην κυρία Κόρχολα καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν μπορούμε να δεχθούμε τη ρουλέτα αυτή που παίζει η Βόρεια Κορέα ούτε και την καταπίεση εις βάρος του λαού της. Την ε, προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύθηκε μια έκθεση η οποία καταδεικνύει ότι έχει επιδεινωθεί η κατάσταση με συνοπτικές εκτελέσεις, υποσυτισμό, στρατόπεδα κράτησης φυλακισμένων σε περιοχές απομονωμένες που καταγράφουν και οι δορυφόροι με 200.000 και πάνω φυλακισμένους που κρατούνται και αξιοποιούνται σε καταναγκαστικά έργα. Η ανθρωπιστική κατάσταση είναι χειρότερη στον κόσμο από ό,τι φαίνεται ή από τις χειρότερες. Αλλά και η αντίληψη της κατάστασης είναι πολύ κακή. Οι κυρώσει που επιβάλλει η διεθνή κοινότητα δεν έχουν καθόλου βελτιώσει την κατάσταση και ελπίζω ότι η πατή εκπρόσωπος κυρία Άστον θα μας πει ποια είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Κύριο Ζέμκιν έχει το λόγο. Πρόεδρε, θα ήθελα να ε, δηλώσω την ευγνωμοσύνη μου για τα όσα ακούστηκαν και έχοντας επισκεφθεί αρκετές φορές ε, τη Βόρεια Κορέα θα θέλω να πω τα εξής υπάρχουν αργά αλλά καθαρά συμπτώματα, ενδείξεις αλλαγής. Κάποιες προσπάθειες, παραδείγματι, που γίνονται για την εισαγωγή του ελεύθερου εμπορίου σε μικρή κλίμακα. Πολυμερείς δράσεις, πιστεύω, μπορούν να φέρουν καλά αποτελέσματα και ίσως είναι καλό να προσέξουμε πολύ τι είδους κυρώσεις θα επιβάλλουμε στην Βόρεια Κορέα. Σε αυτό χρειάζεται να συνεργαστούμε με την Κίνα. Γιατί η Κίνα είναι το μόνο κράτος με το οποίο επιδιώκει να διατηρήσει καλές ε, σχέσεις η Βόρεια Κορέα. Ευχαριστώ. Κυρία Λόχπιλερ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπατή εκπρόσωπε, μας έχει απασχολήσει πολύ και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα και ε, ιδιαίτερα ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τη χαιρετίζουμε και την πρωτοβουλία, να δώσει έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και την θέσπιση μιας ε, ειδική επιτροπής που θα διερευνήσει τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα. Ιδιαίτερα η κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων. 200.000 είναι από ό,τι φαίνεται οι κρατούμενοι για τους οποίους ε, για τους οποίους υπάρχουν καταγγελίες και από αποδείξεις μέσω των καταγραφών σε ε, από που βρίσκονται σε στρατόπεδα κράτησης. Μέσα ναι, αξία αυτών υπάρχουν και παιδιά ακόμη που υποχρεούνται όπως και οι ενήλικες σε καταναγκαστικά έργα. Πρέπει λοιπόν αυτά τα κέντρα κράτησης πολιτικών κρατουμένων, ε, τιμώρησης καλύτερα πολιτικών κρατουμένων, να ε, κλείσουν και να αποφλέξουν όλοι αυτοί. Ευχαριστώ πολύ. Ο Δόκτωρ Τάνοκ έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η Βόρεια Κορέα είναι από τι πιο απομονωμένε και τη δικτατορίε του κόσμου που έχει αποδειθεί και σε πυρηνικό αγώνα δρόμων με δοκιμές πυραυλικών ε, συστημάτων, ενδεχομένως και με πυρηνικές κεφαλές, αποτελεί έναν πολύ μεγάλο κίνδυνο για τη διεθνή κοινότητα. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να την επαναφέρει στην ε, ε, πορεία της υπογραφής της ε, συμφωνίας για την απαγόρευση των όπλων καταστροφής αλλά και προς το δρόμο της συμφιλίωσης με την Νότια Κορέα. Δεν μπορούμε λοιπόν ε, να ξεχνάμε ότι η Ρωσία ακόμη δεν έχει συγχωρήσει τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ προ την Ανατολική Γερμανία που κακώ είχε υποσχεθεί το ΝΑΤΟ ότι θα πράξει. Γι' αυτό και δεν θα είναι καθόλου εύκολο να εξασφαλίσουμε τον αφοπλισμό και τη συμφιλίωση στην ε, Κορεατική Χερσόνησο. Υπάρχει και εκείνη από την άλλη πλευρά. Επομένως θα πρέπει ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή. Κοιτάξτε, θα σταματήσουμε εδώ τη συζήτηση. Ακούγοντα την κυρία Άστον, Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Στην Βόρεια Κορέα βλέπουμε ένα βάναυσο καθεστώς, ένα καθεστώς που ε, κακομεταχειρίζεται φρικτά τους πολίτες του. Το Συμβούλιο των Εθνικών Δικαιωμάτων στην Γενέβη θα κάνει την σχετική διερεύνηση των περιστατικών, αλλά οποιοδήποτε έχει μελετήσει και διαβάσει καταγγελίες όσων μπορούσαν να διαφύγουν από το καθεστώς, γνωρίζει πολύ καλά την τρομοκρατία που επιβάλλει το καθεστώς της Βορειάς Κορέας στους πολίτες του. Επίσης, απλώς, ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα ότι απλώς δεν εξασφαλίζονται τα απαραίτητα για το ζήν στους πολίτες. Το, τρόφιμα, το επιστημικό πρόβλημα είναι τεράστιο για την Κίνα. Έχω συζητήσει με την Κίνα το θέμα της Βόρειας Κορέας στο στρατηγικό διάλογο αρκετές φορές. Προσπαθώ να επισημάνω στην Κίνα το πόσο σημασία θα είχε να υποστηρίξει τη Βόρεια Κορέα σε ένα άνοιγμα. Θα πρέπει να τους ασκήσει μια πίεση βέβαια θα έχει τεράστια σημασία το να ασκήσει η Κίνα πίεση στη Βόρεια Κορέα. Πάντως πρέπει εμείς από πλευρά μας να συνεχίσουμε την άσκηση πιέσεων ε, και να εξασφαλίσουμε ότι θα εκπληρώνουμε τις δικές μας υποχρεώσεις ε, και να μην αφήνουμε στους Βορειοκορεάτες καμιά ε, ψευδέστηση για τις προθέσεις μας. Πρέπει να ασκήσουμε λοιπόν ακόμη πιέσεις. Αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Uh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με εντυπωσιάζει, Πρόεδρε, η ακρίβεια με την οποία ε, διεξάγεται η συζήτηση. Προσέχετε ιδιαίτερο στο χρόνο. Μάλιστα η με ρωτήθηκα νωρίτερα εάν ε, είχα εγώ ζητήσει το λόγο κατά τη διαδικασία του Catch the Eye, αλλά απουσίαζε φαίνεται εκείνη την ώρα και δεν μπόρεσα να μιλήσω. Επομένω, αν μου δίνετε, δώστε την ευκαιρία μετά, στην επόμενη ομιλία. Καλώ, λέει ο Πρόεδρο. Εάν θέλετε, ακόμη και μετά την παρέμβαση τη κυρία Άστον, μπορώ να σα δώσω το λόγο. Αλλιώ θα πρέπει να αλλάξουμε θέμα. Θέλετε το λόγο τώρα. Ναι, Πρόεδρε. Στο επόμενο θέμα θα προτιμούσα να μιλήσω. Το σημειώνουμε για το επόμενο ζήτημα. Κλείνουμε την ε, προηγούμενη συζήτηση. ψηφοφορία θα λάβει, το αγκημένο θα λάβει η χώρα ε, αύριο στις 11.30. Επόμενο σημείο της μέσης διάταξης, εξαιρετικά σημαντικό. Όλα βέβαια είναι σημαντικά, αλλά αυτό ιδιαίτερα. Θα συζητήσουμε με την ε, υπατή εκπρόσωπο το θέμα της Συρίας. Με ειδική αναφορά